Συνάδελφοι, λοιπόν, ξαναρχίζει μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, ξαναρχίζουμε τις συζητήσεις μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Βιτάλ Μορέιρα για τις ε, προσωρινές διατάξεις ε, για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Κύριε Μορέιρα, έχετε τον λόγο. Κύριε Μορέρα, έχετε έξι λεπτά, έτσι το γνωρίζετε. Μπορείτε να τα μοιράσετε και να τα χειριστείτε όπως θέλετε. Κανονικά τέσσερα λεπτά γίνεται για την παρουσίαση του ζητήματος, του θέματος της έκθεσής σας και μπορεί να έχετε δύο για να ολοκληρωθείτε τη συζήτηση. Αν θέλετε να έχετε τρία και τρία ή έξι, όπως θέλετε εσείς θα μπορέσετε εσείς να ε, διαχειριστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας κατά την δική σας διακριτική ευχέρεια. Έχετε τον λόγο λοιπόν κύριε Μορέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, ρυθμίσεις που έχουμε σε σχέση με το ε, διεθνές εμπόριο. Δηλαδή ρυθμίσεις ε, που αφορούν μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της συνθήκης Λισαβόνας. Πράγματι, σε σχέση με την συνέχεια της συνθήκης Λισαβόνας πριν από τρία χρόνια, οι άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις εντάχθηκαν στην εμπορική πολιτική, κοινή εμπορική πολιτική. Και μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστικέ αρμοδιότητε σε σχέση με την κοινή εμπορική πολιτική, αυτό σημαίνει ότι εφ' εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να νομοθετεί και να υιοθετεί διατάξει νομοθετικέ, καθώ επίση και σε σχέση με τι συμφωνίε όσον αφορά τι επενδύσει και ρυθμίσει. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίζουν κάποια πράγματα μόνο αν έχουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν κάποιες, να αναλάβουν κάποιε κάποιες δράσεις. Η συνθήκη της Αβώνας πριν από τρία χρόνια πριν από αυτήν είχαν πολυάριθμες συμφωνίες επενδύσεων με τρίτες χώρες στα κράτη-μέλη. Πάνω από 1.200 τις συμφωνίες. Ο κύριος στόχος αυτών των συμφωνιών είναι, όπως γνωρίζετε, να υπάρχει προστασία σε σχέση με τις αλλοδαπές επενδύσεις έναντι αυθαίρετων δράσεων, για παράδειγμα κατασχέσεων ή άλλων αυθαίρετων δράσεων. Η συνθήκη της Σαββόνας δεν θέσπισε καμιά μεταβατική ρύθμιση ρητή για αυτές τις ήδη ενισχύει συμφωνίες που εφ' εξής θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο μέσα από αυτόν τον κανονισμό να διασφαλίσουμε τη μετάβαση όσο το δυνατόν χωρίς προβλήματα με τις αναγκαίες προσαρμογές σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο όσον αφορά τις ενισχύει ήδη συμφωνίες. Σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό που επί μεγάλο χρονικό διάστημα διαπραγματευτήκαμε το Συμβούλιο, οι διμερείς συμφωνίες που έχουν διαπραγματευτεί μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών πριν από την έναρξη ισχύ της ε, συνθήκης Λισαβόνας συνεχίζουν ε, να υφίστανται ή ε, ας το πω έτσι με την προσαρμογή αυτή μπορούν να καταργηθούν αν αντιβαίνουν διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου ή αν μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλυφθεί δράση εναντίον τους. Επίσης ρυθμίζονται τα πράγματα σε σχέση με τις διμερείς αυτές συμφωνίες μετά από την συμφωνία της Έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Υπό αυστηρού όρου και προϋποθέσεις αυτό ήταν το αντίτιμο το οποίο απέτησε το Ευρωκοινοβούλιο για να νομιμοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες. Και τρίτον, οι όροι και προϋποθέσεις αυστηροί πάντα που τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν ε, την άδεια εφ' να τροποποιήσουν ή να συνάψουν νέες συμφωνίες για τις επενδύσεις σε, περίπτωσεις, περιπτώσεις όπου δεν ενδιαφέρεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί κάτι τέτοιο η ίδια. Το αργότερο μετά από 10 χρόνια θα πρέπει σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνταχθεί έκθεση να εξεταστεί η κατάσταση και να αναλυθεί και να προταθούν οι ε, προσαρμογές και οι αλλαγές που χρειάζονται. Χρειάστηκε λοιπόν μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό και να μπορέσει να είναι πλήρως ικανοποιητική αυτή η συμφωνία και να ανταποκρίνεται στους κυριότερους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς όφελος των συμφερόντων των εταιριών μας και των επενδύσεών μας. Πολύ σας ευχαριστώ Πρόεδρε. <coughs> θα σας απομείνουν δυόμιση λεπτά για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση στο τέλος. Εξ ονόματο τη Επιτροπής έχει τον λόγο κύριος Επίτροπος Κάρεν Χούχτ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου τη Επιτροπής, θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πετύχαμε εξαιρετική συμβαστική λύση στο θέμα αυτό. Διαδοχικοί τριμερής διάλογοι μας επέτρεψαν να εξασφαλίσουμε δημιουργικό επικοδομητικό διάλογο και υψηλή ποιότητα ε, νομοθετικό κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Μορέιρα, για την προσήλωσή τους στην εργασία μας. Ο λόγος για την κατάθεση αυτή τη πρόταση είναι ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα εξυγχρόνισε την κοινή εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δει το θέμα των επενδύσεων που αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο πολιτική. Όλοι συμφωνήσαμε από την αρχή ότι η νέα επενδυτική πολιτική πρέπει να βασίζεται την εμπειρία που έχουμε ήδη αποκομίσει ως κρατημέλη. Οι συμφωνίες επενδύσεων που συνήθισαν τα τελευταία 16 χρόνια αποτελούν πολύτιμο κοινοτικό κεκτημένο. Παρ' όλα αυτά, παράλληλα απαιτείται να καταστρώσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Όπω είπε και ο καθηγητή Μορέιρα, πρόκειται για σημαντικό νομοθετικό κείμενο στον τομέα του εμπορίου, αν και είναι κάτι το οποίο δεν επιτεύχθη εύκολα. Ο τριμερής διάλογος κατέδειξε ότι τα θέματα από θεσμικής και νομικής απόψεως είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Η οριστικοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας, ήδη από την δεύτερη ανάγνωση, πιστεύω ότι θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα για όλους μας. Ο κανονισμός εξασφαλίζει ασφαλεία δικαίου για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Θα συνεχίσουν να εποφελούνται από τις υφισταμένες 1.400 σχετικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες, Έστω του βεβαίω αυτές αντικατασταθούν από συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός περιλαμβάνει όλες τις ε, διασφαλίσεις, βάσει των οποίων δεν θα προκύψουν εμπόδια, σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση τη επενδυτικής μα πολιτική που αποτελεί και σημαντική προτεραιότητα για μα. Η έγκριση λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά τη όργανα να εστιάσουν από εδώ και πέρα την προσοχή του στην υλοποίηση τη επενδυτική μα πολιτική. προωθώντας τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις κατά περίπτωση για να προστατεύσουμε όλους τους Ευρωπαίους επενδυτέ. Σε βάση ισοτιμίας και στο πλαίσιο τη επιτεύξης των στόχων τη εξωτερική μα πολιτικής. Καλό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο του κανονισμού που αφορά τις διμερεί συμφωνίες επενδύσεων. Ω τώρα, ξέρω ότι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου μα υποστήριξε ομοφόνος. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος τώρα των κυλοβρετικών ομάδων θα έχουμε τους αγορητές. Από το ΕΛΚ πρώτα, για δύο λεπτά, η αγαπητή συνάδελφος η κυρία Όμεν Ρόιτεν πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρους του συναδέλφου του κυρίου Σαλάφσκη που είναι τη εισηγητής για την έκθεση αυτή. Ο κύριος Μορέρα τα είπε όλα πολύ καθαρά. Από τότε που ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, οι συμφωνίες για μέρες επενδύσεις είναι μέρος των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι καλό ε, πράγμα ε, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για διμερείς ε, επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα πολύ φοβάμαι. Πολλά κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες που παραμένουν δεσμευτικές όπως λέει αυτός ο κανονισμός. Το ερώτημα όμως είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εξίσου υψηλής ποιότητας ε, όπως οι συμφωνίες που συνήψαν στο παρελθόν τα κράτη-μέλη με τις εν Θα ήθελα να σας απευθύνω μια έκκληση λοιπόν να μην καταλήξουμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή σε σχέση με τις συμφωνίες αυτές, να φροντίσουμε να είναι υψηλής ποιότητας οι συμφωνίες που θα αντικαταστήσουν τις διμερείς. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι το εξή. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν κατάλληλες μορφές διαιτησίας για την ε, διευθέτηση τέτοιων συμφωνιών. Υπάρχει το Διεθνές Κέντρο για επίλυση διαφορών σε θέματα επενδύσεων, βεβαίως. Τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να προσφύγουν σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις και όχι μόνο οι χώρες ε, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιζητήσουν διαιτησία. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να κλείσω θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή έχει διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Η ερώτηση είναι αν η συμφωνία που πρόκειται να συνάψετε με τον Καναδά είναι εξίσου υψηλή ποιότητα ώστε τα κράτη-μέλη να μην χάσουν σαν αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας. Και σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε και πιο δύσκολε χώρε ε, όπω η Κίνα. Θα ήθελα μια απάντηση από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα εξ ονόματο τη Σοσιαλιστική Ομάδα η κυρία Αντρέ Μπαρέα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Όπω έλεγε ο εισηγητή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι οι κανόνε του παιχνιδιού που θεσπίζονται με τι συνθήκε Λισαβόνα σε σχέση και με τις μελλοντικές διμερείς ε, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες και θα πρέπει να θεσπίζονται τα κριτήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να νομοθετούν τα κράτη. Είναι ένα ισόρροπο μέσο αυτό για τα κράτη και να εναρμονιστούν τα πράγματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολο ήταν αυτό διότι είχαν αντισταθεί τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον ας το πω ε, ρόλο που θα τους απέμενε σε σχέση με θέματα διμεριών συμφωνίων συμφωνιών. Όμως ο στόχος είναι να προωθηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις επενδύσεις και να προαθούν οι επενδύσεις και να υπάρχει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Έτσι βρήκαμε τον τρόπο ή ας το πω έτσι τον ακρογωνιαίο λίθο όπως είπε ο Επίτροπος να εγγυηθούμε και να προστατέψουμε τις συμφωνίες των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Να εναρμονίσουμε το πλαίσιο των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό του. Η υλοποίηση, σημαντικό και αυτό, των όρων για την επιδιαιτησία πρέπει να το σημειώσουμε και πρέπει να αναζητούνται στις μελλοντικέ ευθύνε να ζητείτε η οικονομική λογοδοσία και υπευθυνότητα. Αυτό σε χέγγιο και έτσι να μην είναι καταχρηστικές οι συμφωνίες αυτές και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ή αθετήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ Πέπα. Εξ ονόματος των συναδέλφων φιλελευθέρων για δύο λεπτά ο κύριος Ρινάλντι παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η άκρηση αυτή του κανονισμού είναι ένα βήμα πρόοδου σημαντικό προ την κατεύθυνση τη βεβαίωση μια από τι βασικέ αρχέ τη συνθήκη Λισαβόνα, αποκλειστική αρμοδιότητα δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ε, διεθνού εμπορίου. Εκτιμούμε την ε, προσπάθεια που έκανε ο Πρόεδρο Μορέιρα και την συμφωνία που βρέθηκε με το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ε, λυπηρό και πιο αναχρονιστικό από το να παλεύουν μόνα του τα κράτη-μέλη Τη της Ένωσης για να αποσπάσουν την α ή β ε, θετική ρύθμιση μόνο για αυτά τα ίδια. Πιστεύω ότι η Κομισιόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εγγύητης από ό,τι τα επιμέρους κράτη-μέλη για συμφωνίες εγγυητης απο οτι τα επιμέρου κρατη μελη για συμφωνίε πραγματικα ε, ε, χρήσιμες. Είναι πραγματικά λυπηρό και για τη θέση των χωρών μας μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Ε, εδώ στην πρόταση προβλέπεται ένα καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ένα περιθώριο ευελιξία αλλά και επιλύεται μία κακοφωνία. Διότι οι διμερείς αυτές συμφωνίες ε, δεν ήταν μόνο ε, θεμητές ε, ε, εμπορικές συμφωνίες, αλλά και ε, επενδυτικές συμφωνίες, συγγνώμη, αλλά και ένα μέσο ανταγωνισμού μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, διεθνή σκηνή. Πολλά τώρα εξαρτώνται από τη σωστή εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Η Κομισιόν αποκτάει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, ένα ρόλο τον οποίο υποστηρίζουμε ε, πραγματικού εγγυητή της, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όλα τα θέματα που πλέον ε, ρυθμίζονται με πολύ εσωρμένο τρόπο μέσω αυτής της συμφωνίας. Ε, παρακαλώ την Κομισιό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συχνά ε, πλήττονται από τέτοιες επενδυτικές συμφωνίες ενώ ταυτόχρονα είναι το πιο καινοτόμο κομμάτι ε, και το κομμάτι των επιχειρήσεων που δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας στις κοινωνίες μας. Ε, πρέπει να αποδείξουμε ότι η ε, προστασία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αποτελεσματική από αυτή των μεμονωμένων κρατών μελών που ανήκουν σε ένα κόσμο μιας κατακαιρματισμένης Ευρώπης που για μας ανήκει μόνο στο παρελθόν. Ευχαριστούμε για τους πράσινους. Για ένα λεπτό η κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Σκιώδη Συγητή και τον κύριο Ζαλέτσκι για την στεναρή ε, παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας. Οι πράσινοι είμαστε ικανοποιημένοι, μια και το τελικό αποτέλεσμα αφορά τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια νέα πολιτική επενδύσεων. Αυτό ε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση, η ρύθμιση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις νέες αρμοδιότητες. Όμως ο κανονισμός δεν ε, υλοποιεί τον κύριο στόχο του, δηλαδή να μπορέσουν ε, να εκπνεύσουν όλες οι διμερείς συμφωνίες μέσα σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα μεταβατικό και να περάσουμε στο ενιαίο σύστημα. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή στην διαιώνιση αυτών των θεμάτων και δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα ότι κάποτε θα υπάρξει μια τελεσίδικη ρύθμιση και όλα αυτά θα αποτελούν πλέον μια παλιά ιστορία. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι ικανοποιητική λύση σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Δηλαδή την εγγύηση ότι εφ' εξής θα έχουμε μια μεταβατική συμφωνία, προσωρινή συμφωνία για να ρυθμιστούν τα της κοινή πολιτικής για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Gracias. Πρόεδρο, ευχαριστώ Φρανσίσκα. Στη συνέχεια 1,5 λεπτό ο κύριος Πάσκα εξ ονόματος της Ευρώπης των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών που μεταβιβάζονται στην, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οι αρμοδιότητες αυτές συνοδεύονται από διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο της ΕΕ, των κρατών μελών και των εμπορικών εταίρων τους. Εκατοντάδες ε, τέτοιες συμφωνίες που κατά το παρελθόν συνήπταν τα κράτη-μέλη υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς θα πρέπει να καταλήξουν και να ενταχθούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς να υπάρχουν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των συμβαλωμένων μερών. Η αναδιαπραγμάτευση διμερών τέτοιων συμφωνιών ή ε, συμφωνιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά το παρελθόν δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή των προηγουμένων εταίρων. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς θα πρέπει να εξευρεθούν τα πιο σκόπιμα και ενδεδειγμένα μέτρα και ε, πολιτικές μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας. Με τη νέα διαπραγμάτευση θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της ενημέρωσης και μία από τις δυνατότητες που τεχνικά και οργανωτικά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την περίπλοκη δηλαδή διαδικασία μια τέτοια δυνατότητα θα είναι η μεταφορά των ε, εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετάθεση αυτών των ε, εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συνάδει σε σχέση με τον κανονισμό 182-2011. Και ως προς ε, όλα αυτά μια και πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκες διεργασίες θα πρέπει να μπορέσουμε να εργαστούμε με τον ακριβέστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκο. Ολοκληρώσαμε αυτό το γύρο. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων και για 1,5 λεπτό ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν έχει το λόγο. I. ήταν αυτό το οποίο έφερε στο τέλος ε, της προηγούμενης χιλιετίας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο για να διαδηλώσουν. Η λεγόμενη πολυμερή συμφωνία επενδύσεων και στόχο είχε να διασφαλίζει τις μεγάλες εταιρείες παγκοσμίω κατά οποιασδήποτε μορφής ε, επέμβασης ε, των τότε ακόμα κυρίαρχων κρατών. Οποιαδήποτε μορφή ε, κρατικοποίησης ήταν αδύνατη. Περιορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ανταυτού καταλήξαμε στην πάρα πολύ γρήγορη ε, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί επειδή αποτύχαμε σε αυτό, επειδή ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους, λένε τουλάχιστον ας σιγουρέψουμε τη διεύρυνση. Παράλληλα με αυτό αναπτύχθηκαν οι διμερείς συμφωνίες. Και τώρα συνοψίζονται όλα αυτά επί της αρχής. Εάν κάποιος ε, όπως εγώ είναι υπέρ της Ευρώπης αλλά κατά αυτών των ακραίων συμπεριφορών, το ερώτημα είναι ουσιαστικά τι γίνεται. Τι γίνεται με τα διπλώματα βρεστεχνία, τι γίνεται με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι κάνουμε με τι χώρε τη Αφρική. Εάν δηλαδή ε, υπάρχει η απαραίτητη προστασία και των ε, αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και των δικών μας εταιριών και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει από κάποια άλλη αφετηρία αντί για να σκέφτε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μετά από τις ομάδες, θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι με μεμονωμένα. Ο κύριος Σαλεύσκη έχει το λόγο για δύο λεπτά καταρχήν. E, e, είναι ε, ένας πολύ σημαντικός αυτός ο κανονισμό που θα ψηφίσουμε αύριο στην Ολομέλεια επειδή δείχνει πώ αυτό το σημαντικό στοιχείο τη συνθήκης για την κοινή επενδυτική πολιτική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μεταξύ των σοσιαλιστών φιλελευθέρων μελών του ECR και τον Επίτροπο Ντεγκούχτ του οποίου η ομάδα εργασίας πρότεινε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Οι πράσινοι πρότειναν μια πολύ, έναν πολύ ενδιαφέροντα κοινό κανονισμό ο οποίος μεταφέρει το βάρος της προστασίας των συμφερόντων των Ευρωπαίων επενδυτών ε, στην ε, ευρωπαϊκή πλευρά. Ο κανονισμός που θα ψηφίσουμε αύριο είναι επίσης κοινή κοινοτική πρόταση. Δεν προχωράει τόσο μακριά όσο η πρόταση των πρασίνων συναδέλφων, αλλά ο κανονισμός αυτός εμπεριέχει τους πιο σημαντικούς κανόνες. Πρώτα, ένα σύστημα προστασίας των Ευρωπαίων επενδυτών κοινό Όλοι θα προστατεύονται δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι κάποιες χώρες εποφελούνται από τα διαφορετικά επίπεδα εγγύησεων για να ασκήσουν πολιτική πίεση σε κάποια από τα κράτη-μέλη μας και όσο του καταλήξουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας οι τρέχουσες, ε, θα ισχύουν οι τρέχουσες συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατό θα παίξει σε αυτό σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι του χρόνου θα έχουμε μια πρώτη συμφωνία με τον Καναδά και τις δικές μας κοινοτικέ συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το στάδιο όταν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, τα δικά μας ε, συμφέροντα, τα κοινοτικά συμφέροντα είναι αυτά που πρέπει να επικρατήσουν. Έληξε ο χρόνος σας. Για ένα λεπτό έχει το λό. Ο κύριος Ζαν Ευχαριστώ πρόεδρε. Αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζω να μπορέσει να εκφραστεί θετικά επί του κανονισμού αυτού που αποτελεί βασικό στοιχείο συνδρομή στην εμπορική πολιτική με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βιντάλ Μορέιρα και την Επιτροπή του που πρόθυσε αυτό το ζήτημα προωθούμε θέματα της συνθήκης γιατί δεν υπάρχει κατακαιρματισμός ε, των επενδυτικών συμφωνιών και όπως είπε και ο συνάδελφος Ρινάλτη δεν γίνεται εσωτερικό ε, dumping μεταξύ των 27 ε, κρατών μελών ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των επενδυτικών μέσων. Άρα μιλάμε για ασφάλεια επενδύσεων, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας που και το μεταβατικό καθεστώς. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν για την εμπορική μας ε, πολιτική γενικότερα. Ευχαριστούμε. Ο γύρος αυτός θα κλείσει με τον κύριο Αντρέα Μέλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τις ε, συνθήκες ε, της ε, φιλίας και της ναυτιλίας των προηγουμένων δεκαετιών και αιώνων οδηγηθήκαμε στις τωρινές συμφωνίες και έχουμε καταλήξει σε ένα σύστημα το οποίο πλέον είναι ακατανόητο. Έχουμε φοβερές, φοβερό περιορισμό του ρυθμιστικού ρόλου του κάθε κράτους και έχουμε εταιρείες τον οποίο ο τζίρος ξεπερνάει το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών και μπόρεσαν να αναπτυχθούν ακριβώς μέσω αυτών των συμφωνιών. Και βεβαίως υπάρχει και ο ρόλος των νομικών στις διάφορες αυτές ρήτρες προστασίας των επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, αντιβαίνει τις ίδιες τις, τις πολιτικές μέσω ακριβώς αυτών των συμφωνιών για εγγυήσεις εξαγωγών και προστασίες επενδύσεων καθώς αυτές έχουν φοβερές συνέπειες ως γνωστόν για τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα πρέπει να βρεθούν και λύσεις στις ε, περιπτώσεις εκείνες ε, στις οποίες απειλείται ένα κράτος μέλος όταν παραβιάζει μια τέτοια συμφωνία για κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, είχαμε κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες μεταβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν πριν υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία με την Κίνα. Έχουμε δύο συναδέλφους που ζητούν ε, να παρέμβουν βάσει βάση το Catch the Eye. Η κυρία Τσικάου καταρχήν. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζουμε τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου για τα μεταβατικά ε, μέτρα σε σχέση με τις επενδυτικές συμφωνίες ε, μεταξύ κρατών μελών. Δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη έχουν διαπραγματευτεί και συνάψει διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε άμεσες επενδύσεις. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ορίζουμε ένα πλαίσιο και τους όρους ε, δυνάμει των οποίων μπορούμε να αλλάξουμε μία διμερή συμφωνία. Έτσι τα κράτη-μέλη θα, θα μπορέσουν να ε, συνάψουν συμφωνίες, νέες διμερείς ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε. Κλείνει αυτός ο γύρος με τον κύριο Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την συνθήκη της ε, Λισαβόνας πλέον οι άμεσες ε, ξένες επενδύσεις ανήκουν ε, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να κλείσουν τέτοιες συμφωνίες εάν τις εξουσιοδοτήσει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι περιορίζονται πάρα πολύ τα δικαιώματα των καρτών μελών και υπάρχουν προβλήματα με την νομική ασφάλεια δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά για επενδυτές από την Ένωση να ισχύουν οι υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας. Εάν είναι οι συμφωνίες ενός κράτους μέλους με υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει αυτές να ισχύουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε με τις παρεμβάσεις και θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος για να απαντήσει στις διαφορές παρεμβάσεις. Έχετε το λόγο κύριε Ντεχούχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αντιδράσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν στη διάρκεια αυτής της συζήτησης η οποία έδειξε ότι υπάρχει γενικά υποστήριξη για την πρόταση που έχουμε υποβάλει μέσα από τις διαπραγματεύσεις, το τριμερή διάλογο υπό την εποπτεία του καθηγητή Μορέρα με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο κείμενο το οποίο σας έχουμε υποβάλει. Η κυρία Ράιτεν έθεσε μία ερώτηση ρωτώντας θα έχετε το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας που υπάρχουν σε διμερείς ε, συμβάσεις ε, χρηματοδότησης αυτό, ε, και επενδύσεων. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι κάθε κράτος μέλος θα εξασφαλίσει την ίδια υψηλή προστασία που αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για λίγες χώρες. Να δούμε τις ε, συνθήκες σε ορισμένες χώρες. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένες Πρέπει βεβαίω να δούμε και ποιο είναι το μέγεθο, η έκταση αυτού του κράτου μέλου. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε κράτο μέλο, ακόμα και τα πιο μικρά, θα απολαμβάνουν του ίδιου υψηλού επίπεδου προστασία που επιφυλάσσεται, που αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για ε, μια ή δυο χώρε σε κάποιε περιπτώσει. Δεύτερον, θα δημιουργήσει αυτό ε, κάποιο εσωτερικό σύστημα. Δεν το νομίζω. Έχουμε ζητήσει την διαπραγμάτευση ε, διαφόρων ε, ε, εντολή για τη διαπραγμάτευση τέτοιων συνθήκων επενδυτικών συνθήκων με διάφορες χώρες όπως η Ινδία παραδείγματος χάρη και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το Συμβούλιο μετά από τη σχετική συζήτηση αλλά μας έδωσαν την εξουσιοδότηση να διαπραγματευτούμε εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, είναι, θα, καταργηθεί στο, σταδιακά. Όχι, διότι τα κράτη-μέλη όλο και περισσότερο θα επιμένουν αυτές οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες να αποκτήσουν ευρωπαϊκή εμβέλεια, να γίνουν ευρωπαϊκές επενδυτικές συμφωνίες. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε την ίδια προστασία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι εκείνα που θα επιμείνουν να ε, ε, από τις διμερείς επενδυτικές ε, συμφωνίες να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκές ε, ε, επενδυτικές συμφωνίες και γι' αυτό συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απομακρυνθεί από την αρχική της πρόταση για την μείωση της σταδιακής κατάργησης μετά από κάποιο διάστημα. Ε, μετά από όριμη σκέψη, η δυναμική των κρατών μελών που θέλουν το ίδιο επίπεδο προστασίας είναι αυτή που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ταυτόσιμο για όλα τα κράτη-μέλη και αυτό ε, είναι ε, είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο για τον εισηγητή αλλά και για την Επιτροπή ε, να μπορέσουμε να συναντηθούμε με έναν επίτροπο που γνωρίζει το θέμα και δεν έρχεται απλώς για να μας διαβάσει ένα χαρτί. Ε, εκτιμούμε την παρουσία όλων βεβαίως και γνωρίζετε ότι ε, ε, θεωρούμε ότι ο συνομιλητής μας θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το θέμα που μας απασχολεί. Έτσι βελτιωνόμαστε και εμείς. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Βιτάλ Μορέιρα, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επενέσω τον κύριο Ντεχούχτ για τις γνώσεις του και μπόρεσε να ανταποκριθεί στα, σε όλα του τα επιμέρους καθήκοντα και φακέλους παρά το άτυχο τέλος της άκτα. Επρόκειτο για μια διαπραγμάτευση που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Θεωρήσαμε ότι η διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να είναι επίσης αποκλειστική μας αρμοδιότητα. Και υπάρχει και προστιθέμενη αξία με βάση μια κοινή πολιτική, πολιτική εξωτερικού εμπορίου παρά να έχουμε μια κατακαιρματισμένη πολιτική 27 κρατών μελών. Στο τέλος αυτής της δύσκολης διαπραγμάτευσης θα πρέπει να τονίσουμε την σοβαρότητα και τη δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων. Χωρίς ε, την Πολωνική Προεδρία και την ε, Δανική δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καταλήξει. Επίσης, ε, χωρίς την συνεισφορά της Κομισιόν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε συμφωνία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Ζωακίμ Μασάδο, τον ρόλο του Ζωακίμ Μασάδο ο οποίος μπόρεσε να οδηγήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις σε αίσιο πέρας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, Πάβελ Ζαλεύσκη, ο οποίος δεν, δεν αποδυνάμωσε το κείμενο. Άρα πιστεύω ότι θα ψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο βήμα για την ε, σωστή προώθηση του εξωτερικού μας εμπορίου. Νομίζω ότι θα είμαστε μία πιο ε, θα έχουμε πιο στενές σχέσεις με όλους τους εταίρους στο εξωτερικό εμπόριο. Ευχαριστούμε Βιτάλ. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια έχουμε άλλη μια έκθεση του Βιτάλ Μορέιρα, μακροοικονομική χρηματοδοτική σύνδεση.